για την προστασία των συμφερόντων των τοπικών πιστωτών. Τέταρτον, η πρόταση απαιτεί από τα κράτη-μέλη να δημοσιεύουν τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις σε διασυνοριακές υποθέσεις αφαιρεγγιότητος, σε ηλεκτρονικό μητρό, προσπελάσιμο από το κοινό και προβλέπει τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων αφαιρεγγιότητας. Επίσης προβλέπει τυποποιημένα έντυπα για την αναγγελία των απαιτήσεων. Και πέμπτον, η πρόταση προβλέπει συντονισμό των διαδικασιών αφαιρεγγιότητος που αφορούν διαφορετικά μέλη του ίδιου ομίλου εταιριών, υποχρεώνοντας τους συνδίκους και τα δικαστήρια που εμπλέκονται στις διαφορές να συνεργάζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον Ιουνίου του 2013 πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συζήτηση προς ανατολισμού και υιοθετήθηκαν κάποιες προτινόμενες γενικές κατευθύνσεις, κατευθυντήριες γραμμές για το μελλοντικό έργο της ομάδας εργασίας. Αυτές συνίστανται σε επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε προπτωχευτικό στάδιο, παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε βιώσιμες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες φυσικά πρόσωπα. Δεύτερον, στη δικαιοδοσία για το άνοιγμα διαδικασιών αφαιρεγγιότητος, γίνεται δηλαδή αποσαφήνιση της έννοιας του κέντρου των κυρίων συμφερόντων για την ε, θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας με κριτήρια που θα αποτρέπουν την άγρα δικαστηρίων. Και ε, δημιουργία, γίνεται δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου αφαιρεγγιότητος σε όλα τα κράτη-μέλη με διασύνδεση μεταξύ τους και με πρόσβαση σε αυτά μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση εφερεγγιότητας εταιριών μελών ομίλων επιχειρήσεων και γίνεται μια όσο το δυνατόν πιο σύντομη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί του κανονισμού σύμφωνα και με σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ελληνική Προεδρία αναγνωρίζει τη σποδιότητα της πρότασης κανονισμού όσον αφορά τον τομέα δικαιοσύνη για την ανάπτυξη και συμφωνεί πως ο εξυγχρονισμός των κανόνων περί αφαιρεγγιότητος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διευκολύνει μεταξύ άλλων τη διάσωση και την αποκατάσταση των βιώσιμων επιχειρήσεων ώστε οι επιχειρηματίες να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη σημαντική πρόοδο των εργασιών για την τροποποίηση του κανονισμού περί με επιθυμητό σκοπό την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Ως προς την πρόταση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πολίσεων. Η Ελληνική Προεδρία αναγνωρίζει τη σημασία της πρότασης κανονισμού για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων. Είναι κατανοητό ότι μέσω ενός τέτοιου κειμένου προάγεται η εναρμόνιση ενός ουσιαστικού τμήματος του αστικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς και της ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντων. Η πρόταση προβλέπει τη θέσπιση κοινού, ευρωπαϊκού δικαίου των πολίσεων και εναρμονίζει τα εθνικά δίκαια των συμβάσεων των κρατών μελών με την καθιέρωση εντός του πλαισίου του εθνικού δικαίου εκάστου κράτου μέλους ενός δεύτερου καθεστώτος δικαίου των συμβάσεων για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, το οποίο θα είναι πανομοιότυπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεπάρχει με τους προϋπάρχοντες κανόνες του εθνικού δικαίου των συμβάσεων. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων θα είναι εφαρμοστέο προαιρετικά στην εκάστοτη διασυνοριακή σύμβαση έπειτα από σχετική ρητή συμφωνία των συμβαλωμένων μερών. Γνωρίζουμε ότι εκτός από τις αντιδράσεις κρατών μελών στο Συμβούλιο, διαφορετικές θέσεις έχουν σημειωθεί και στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζουμε επίσης ότι η Επιτροπή σας υιοθέτησε έκθεση με την οποία μάλιστα ζητεί την τροποποίηση πολλών άρθρων καθώς και τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής αποκλειστικά στις εξαποστάσεως πωλήσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε τη συζήτηση και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο τέλος Φεβρουαρίου. Η Ελληνική Προεδρία, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που εντοπίζονται κατά την επεξεργασία του νομικού αυτού εργαλείου, θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της επικοδηματικής συνέχισης των διαπραγματεύσεων του νομοθετήματος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σα ευχαριστώ θερμά κύριε Υπουργέ. Θα έλεγα είναι τρεις σημαντικότατοι άξονες αυτοί που προαναφέρατε. Και υπάρχει εδώ κάπως το κόλλημα ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ελληνικής προεδρίας, ναι με το, ε, την έχουμε κατά το πρώτο εξάμεινο που είναι προτέρημα, από πλευράς ε, χρονικής. Όμως τον Απρίλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον τέταρτο μήνα θα σταματήσει τις δραστηριότητες του λόγω ευρωεκλογών. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι ε, έχει συνμηθεί ο χρόνος ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ολοκλήρωση με την Ελληνική Προεδρία. Δυστυχώς όμως αυτό συμβαίνει με το χρονοδιάγραμμα από χρονικής πλευράς. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι επικεντρώνεστε σε αυτούς τους τρεις κυριότερους άξονες. Διότι πράγματι είναι πολύ σημαντικοί αυτοί οι άξονες Τώρα ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Πρώτος η κυρία Λίχτενμπεργκερ. Παρακαλώ. Πρώτη κυρία Λίχτενμπεργκερ. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Υπουργέ για το ότι είσαστε παρόν και προσήλθατε εδώ. Μία ερώτηση θέλω να θέσω όπου δυστυχώς την απάντηση δεν θα μπορέσω να παραμείνω να την ακούσω. Έχω παράλληλα μια άλλη κοινοβουλευτική ε, επιτροπή και πρέπει να πάω σε εκείνη. Όμως ε, θέλω να την θέσω την ερώτηση και οι συνάδελφοι θα μου διαβιβάσουν την απάντησή σας οπωσδήποτε. Ένα θέμα να θίξω και να ερωτήσω που τώρα θα μπορούσε να ολοκληρωθεί οπωσδήποτε. Και εδώ πρόκειται Πρόκειται λέγω για ένα ζήτημα για την προσχώρηση οκτώ κρατών στη Σύμβαση της Χάγης για την αφαίρεση παιδιών, απαγωγή παιδιών που μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφενός και του Συμβουλίου αφετέρου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για αυτό το θέμα και την αντιμετώπιση του όσον αφορά τις αρμοδιότητες. Αυτό που οδηγεί. Οδηγεί η διαδικασία αυτή να έχει ξεκινήσει αλλά τώρα να βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο, να έχει αποτελματωθεί η υπόθεση αυτή. Βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. Γιατί? Διότι το Συμβούλιο την περαιτέρω επεξεργασία και εκπόνηση αυτού του θέματος από το Ευρωκοινοβούλιο δεν την εγκρίνει δεν την εγκρίνει. Αυτό τι έχει σαν επίπτωση. Οχτώ χώρε. μεταξύ αυτών και η Ρωσία για παράδειγμα και βορειοαφρικανικά κράτη όπω το Μαρόκο μεταξύ αυτών όπου εδώ και μεγάλο, μεγάλο χρονικό διάστημα επιθυμούμε και ελπίζουμε να προσυπογράψουν αυτή τη σύμβαση, αυτή τη συνθήκη, διότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που εκκρεμούν και θα έπρεπε να διευθετηθούν, να διεκπαιρεωθούν. Όλα αυτά έχουν παγώσει και βρίσκονται αποτελματωμένα όλα. Και θα ήταν λοιπόν πραγματικά ευκταίο γιατί Πρέπει κάποτε να ξεφύγουμε, να διαφύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Πρέπει να εξευρεθεί μια λύση λοιπόν. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Το Συμβούλιο θα μπορούσε να δώσει την άδειά του, την έγκρισή του, να συνεχιστεί η εξέταση και διεκπαιρέωση αυτού του θέματος. Διότι δεν θα μπορέσουμε διαφορετικά θεωρητικά να επιλύσουμε αυτό το θέμα ε, μόνο θεωρητικά κατά το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει λοιπόν εδώ οπωσδήποτε να εξευρεθεί μια λύση προ όφελο και συμφέρον των πολιτών. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση προ εμά κύριε Υπουργέ κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου. Επιτέλους να μεριμνήσετε εσείς ώστε αυτή η διαδικασία να συνεχιστεί. Εδώ πραγματικά πρόκειται για την ευημερία, την ε, ευημερία των γονιών και των παιδιών που βρίσκονται ούτως ή άλλως σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση διότι έχουν χωριστεί τα μέλη αυτών των οικογενειών το ένα από το άλλο και η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να επιδεινωθεί ακόμα περαιτέρω να ζουν αυτοί οι άνθρωποι σε μια θεά νομική ζώνη. Έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο η Ευρώπη αυτές τις 8 χώρες να τις πείσει να κινηθούν ώστε να υπάρξει λύση, να υπάρξει δυνατότητα συνεννοήσεων ενετικών λύσεων. Δεν είναι όμως κάποια αρμοδιότητα, δεν ε, υπάρχει οποιαδήποτε, ας το πω έτσι, ξεχωριστή κατάσταση για τις αρμοδιότητες ή ουδήποτε, όμως έχει χειροπιαστά αποτελέσματα για τη ζωή πολλών ανθρώπων. Θα χαιρόμουν αν μπορούσατε να καταβάλλετε προσπάθεια υπέρ αυτών. Σας ευχαριστώ. Εσείς συνάδελφοι έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον κύριο Υπουργό για αυτές τις πραγματικά διαφωτιστικές και ευσύνοπτες πληροφορίες και για το ότι υποσχεθήκατε σε αυτό το διάστημα όχι να υποβάλλετε ένα ευρύ κατάλογο ως ευχολόγιο για διάφορα θέματα, αλλά να επικεντρωθείτε σε ουσιώδη θέματα, σε σημαντικούς άξονες και αυτό είναι πολύ θετικό το ε, τα νομικά μέσα και εργαλεία για την οικονομική ανάπτυξη να μπορέσουν να επηρεαστούν για την ενιαία εσωτερική αγορά, την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά. Έχω υπόψη εδώ τις ρυθμίσεις για παράδειγμα για το το δικαίωμα για τις πωλήσει ε, και τις ρυθμίσεις για τα θέματα συναλλαγών και πωλήσεων ή την ε, αντιμετώπιση πτωχεύσεων και την αντιμετώπιση αφαιρεγγιότητας. Πώς βλέπετε τις ευκαιρίες αυτά τα θέματα να μπορέσουν πριν από την ολοκλήρωση της δικής σας προεδρίας να μπορέσουν να οριμάσουν και να ολοκληρωθούν. Και ρωτώ και με κάποια ανησυχία. Δεν είναι πρόβλημα της ελληνικής προεδρίας αλλά είναι και της επόμενης προεδρίας. Ε, διαδόχου προεδρίας. Προτού ξεκινήσει το επόμενο νέο εκλεγέν κοινοβούλιο θα έχουμε και το θέμα της εκλογής ε, των, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνέχεια μήνες ολόκληροι θα περάσουν μέχρι να διευθετηθούν όλα αυτά. Είναι κατακαιρματισμός ε, του κοινοβουλευτικού έργου έργου. Πώς μπορεί να επηρεαστεί λοιπόν θετικά η οικονομική ανάπτυξη. Να πάμε με τέτοιο τρόπο να προχωρήσουμε ώστε να ευδοκιμήσουν οι προσπάθειες αυτές. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το εγχείρημα να ληφθεί υπόψη και να μπορέσει να προαχθεί. Και για να υπάρξει και μια προστασία, ας το προσθέσω και αυτό, ε, σε σχέση με οποιασδήποτε αναταράξεις ε, για την Ευρωπαϊκή Ενιαία Εσωτερική Αγορά. Και κατά δεύτερο λόγο σας ευχαριστώ θερμά κύριε Υπουργέ προσωπικά για την ήδη θετική συνεργασία όσον αφορά την φάση Βρυξελών 1. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και ε, διάλογο που θα ε, συνεχιστεί και όταν ε, θα πρόκειται για την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά πράγματα θα είμαστε μετά στη συνέχεια να διασφαλίσουμε μια ομαλή λειτουργία και για το ενιαίο ε, δίπλωμα ε, ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Σας ευχαριστώ. Εσείς συνάδελφε έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν σας εύχομαι κάθε επιτυχία κυρία Θανασίου κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στο έργο σας. Για τα θέματα τα οποία με θετικό τρόπο και σαφήνεια θέσατε στο επίκεντρο θέλω να πω ότι φυσικά θα έχετε την πλήρη υποστήριξη των Ευρωβουλευτών από πλευράς μας. Θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε να υπάρξει χειροπιαστό αποτέλεσμα και για τις πτωχεύσεις και για την ε, αντιμετώπιση της αφαιρεγγιότητας, μια και τα αναφέρατε αυτά. Θα ήθελα όμως να θέσω και στα πρακτικά πρόταση εδώ και κίνητρο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο τον εναρμονισμό για τα θέματα αφαιρεγγιότητας αλλά και για τις πτωχεύσεις ε, και για τις ιδιωτικές ε, αυτές ε, χρεοκοπίες ή πτωχεύσεις όπως στην Ισπανία για παράδειγμα που έχασαν χιλιάδες ή μυριάδες κιόλας πολιτών της Ισπανίας τα διαμερίσματά τους, τα σπίτια τους. Ερώτηση δική μου προς εμάς κύριε Υπουργέ. Στην Ολομέλεια είχαμε με την έκθεση για την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια για την εκπροσώπηση των γυναικών εκεί. Υπήρξε μεγάλη συνένεση. Η συγγήτρια από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας ήταν η συνάδελφός μας από την Ελλάδα Ρόδη Κράτσα. Ερώτησή μου προς εμάς Υπουργέ. Υπάρχει κάποια ευκαιρία για αυτό το θέμα η Ελληνική Προεδρία να επιληφθεί αυτού του θέματος και να οδηγήσει στο να ολοκληρωθεί. Κατά πόσον βρίσκεστε σε στενή συνεργασία ε, σας αναφέρω αυτό άμεσα προς εμάς με τους συναδέλφους σας που έχουν ιδιαίτερες επιφυλάξεις ίσως για αυτό το θέμα. Πώς μπορείτε εσείς να επηρεάσετε αυτό το θέμα και ποιες προοπτικές βλέπετε να υπάρχουν. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το θέμα της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Και είσαστε επαγγελματίας και γνωρίζετε τα θέματα και πραγματικά τώρα συνειδητοποιούμε ότι αυτό το θέμα έχει τεράστια εμβέλεια και βρίσκεται ακόμα στα σπάργανα. Όμως όπως το χρονοδιάγραμμα πρόγραμμα από ό,τι άκουσα από εσά, μια και είναι δεδομένο, από πλευρά ε, του Συμβουλίου θα υπάρχει σίγουρα κάποιο συμφέρον να σημειωθεί πρόοδο και να προχωρήσει αυτό το χαρτοφυλάκιο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με ενδιαφέρει να ακούσω κατά πόσον είναι ένα θέμα αυτό που με μεγαλύτερη προώθηση, με μεγαλύτερη προαγωγή θα δίνατε κάποιε προσπάθειε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μασεπίνταλγο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχηθώ και εγώ ό,τι καλύτερο, διότι γνωρίζω τη χώρα σας συμπάσχω με την κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο. Μου δημιούργησε κάποια αίσθηση νοσταλγίας όταν η κυρία Ποδηματά άκουσε κάποιον ευρωβουλευτή να μιλά από τα ελληνικά εγώ ως νέος μάθαινα αρχαία ελληνικά, έκανα και μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά, κάτι το οποίο φυσικά μάλλον σήμερα δεν θα μπορώ να κάνω, τουλάχιστον όχι όσο θα ήθελα, απλώς και μόνο για να θυμηθώ υπέροχα κείμενα της ε, ε, ελληνικής γλώσσας. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω μια ερώτηση, η οποία μπορεί ίσως να θεωρηθεί άκερη, αλλά είναι και κάπως ευαίσθητη. Προς το τέλος της Λιθουανικής Προεδρίας, η ελληνική αντιπροσωπεία ε, επισκέφθηκε τους σκιώδεις εισηγητές ε, για την οδηγία και τον κανονισμό για τους οικονομικούς ελέγχους ε, και ε, ζητήσαμε να υπάρχει κάποιος πολιτικός ρολισμό ως και αυτό το οποίο καταφέραμε να έχουμε σήμερα το πρωί στην ε, ψηφοφορία που κάναμε για τους οικονομικούς ελέγχους ε, και από τα αποτελέσματα του Συμβουλίου είχε διαφανεί ότι τα πάντα πήγαιναν μια χαρά ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα είτε στην πρώτη ολομέλεια του Φεβρουαρίου είτε στη δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου το αργότερο το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Σήμερα το πρωί όμως μου είπανε ότι τα χόρταγα λόμπι των μεγάλων τεσσάρων εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιημένοι. Ακόμα και αν εμείς να είμαστε ικανοποιημένοι, αυτοί λοιπόν είναι δυσαρεστημένοι και θέλουν να παρακολύσουν ε, και άλλο την έγκριση ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτών των κειμένων που ήδη έχουν συμφωνηθεί μέσω των τριμερών διαλόγων. Θα ήθελα λοιπόν Ε, το γεγονό ότι δεν το αναφέρατε να μην σημαίνει τίποτα, Απλώ θα ήθελα να διασφαλίσω ότι δεν θα δεχτείτε οποιοδήποτε ανάχωμα στην όλη αυτή διαδικασία, ώστε αυτά τα νέα κείμενα τα οποία δεν με ικανοποιούν απόλυτα μεν αλλά και τα καταψήφισα κιόλα, αλλά θεωρώ ότι δεν θα ήταν σωστή ε, πρακτική να δεχτούμε τι πιέσει αυτών των επωνίδιστων ε, λόμπι που προσπαθούν να παρακολουθήσουν το έργο μα. Ευχαριστώ, δεν ζητούν άλλοι τον λόγο. Ούτε και εσεί Ωραία. Τότε λοιπόν ο κύριος Υπουργό θα λάβει τον λόγο. Ε, Α, κυρία Βίξτρομ πρώτα. Συγγνώμη, κυρία Βίξτρομ, παρακαλώ. σα ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια πίεση που δημιουργήθηκε, γι' αυτό ε, και όλα συζήτησα να παρέμβω. Έχω την εντύπωση ότι μπορώ να και πρέπει να πω κάτι. Λοιπόν, εντάξει. Εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο πάντα ασχολούμαστε με τα δικαιώματα των γυναικών και η προλαλή σας συνάδελφο το ανέφερε και κάναμε αυτή τη δουλειά και πριν από κάποια χρόνια είχαμε και κάποια, α το πω έτσι, ε, εξετάσει και τη δυνατότητα απαγορεύσεων. Δηλαδή, αν μια γυναίκα ταξιδεύει σε μια άλλη χώρα, σύζυγος να μπορεί να έχει δικαίωμα επίσκεψης. Αυτό είναι και το δικαίωμα της ελευθερίας κυκλοφορίας που κάθε Ευρωπαίος πολίτης απολαμβάνει αυτών των ελευθεριών. Είναι σαφές ότι οι γυναίκες πρέπει ελεύθερα να μπορούν να κυκλοφορούν. Όμως υπάρχει, ε, επισκιάζεται το θέμα αυτό διότι διαδραματίζει κάποιο ρόλο που και πώς μπορεί να μετακινηθεί μια γυναίκα σε σχέση με τα όσα επιθυμεί ο σύζυγός της κατά πόσο θα σας εσείς πρόθυμος να σημειωθεί πρόοδος ε, σε αυτό το θέμα για αυτές τις δυνατότητες και καλά, καλό είναι ότι υπάρχουν, να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και ελπίζω και πιστεύω ότι η Ελληνική Προεδρία θα καταβάλει προσπάθειες ώστε να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρωτοβουλία όπως ε, το έθεσε στο θεματολόγιο της, στην ημερήσια διάταξή της. Θα ευχόμαστε όλοι και θα χρωστούσαμε ευχαριστίες στην Ελλάδα αν μέσα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας πραγματικά αυτές οι προσδοκίες θα μπορούσαν να αποκτήσουν σάρκα και οστά. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε κυρία Βίξτρομ, κύριε Υπουργέ και τον λόγο. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για τις ε, ερωτήσεις και τις υποκαταενότητες. Ε, όσον αφορά το θέμα της απαγωγής των παιδιών, ε, έφυγε η συνάδελφος που ρώτησε λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις της κυρίας Εναντέλφου και θα προσπαθούσαμε να δούμε τι λύση μπορεί να δοθεί στο ζήτημα αυτό. Πρέπει όμως ε, νομίζω να περιμένουμε και την απόφαση του δικαστηρίου, την απόφαση δηλαδή στην οποία προσέφυγε η Επιτροπή. Να δούμε τι απόφαση θα εκδοθεί. Τώρα, για το θέμα της ε, αφαιρεγγιότητας πράγματι θα βοηθήσει την ανάπτυξη της αγοράς και των ε, ε, των συναλλαγών. Πρέπει να σας πω ότι η εφαρμογή για, επί 13 περίπου έτη του κανονισμού 1346, ήταν ο προηγούμενος κανονισμός του 2000 για την αφαιρεγγιότητα, έχει αναδείξει τα σημαντικά πλεονεκτήματα και την συνεισφορά του κανονισμού αυτού στο διασυνοριακό επίπεδο των πτωχεύσεων. Παράλληλα όμως ανέδειξε και ορισμένες αδυναμίες και δυσλειτουργίες, ιδίως στη δευτερεύουσα διαδικασία πτώχευσης σε ζητήματα αφαιρεγγιότητος, ομίλων επιχειρήσεων και στις προπτωχευτικές διαδικασίες. Αυτές τις ανδυναμίες έρχεται να καλύψει τώρα ο νέος κανονισμός, έτσι ώστε το σύστημα της αφαιρεγγιότητας σε διασυνοριακό επίπεδο να γίνει πιο αποδοτικό και πιο αποτελεσματικό προς όφελος των κρατών μελών ε, και της ίδιας βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας και κατά επέκταση της οικονομίας. Τώρα στο θέμα το δικαίωμα της επίσκεψης των γυναικών είναι, εμείς ε, το βλέπουμε θετικά, είναι σωστή η παρέμβασή σας, είναι αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών όπου υπάρχει και ειδική γραμματεία ισότητος των φύλων και είναι στην άλλη επιτροπή ο κύριος ε, Μιχελάκης. Θα το θέσω όμως ε, υπόψη του, οπότε θα ελπίζω να σας δοθεί και απάντηση σύντομα. Πάντως ε, θετικά αντιμετωπίζεται ότι πρέπει να υπάρχει μια, ε, το δικαίωμα επίσκεψης διότι βοηθά και στην κατά κάποιον τρόπο αν όχι μόνιμη μια επανένωση των, ε, των οικογενειών και είναι, είναι θετικό. Τώρα για τους οικονομικούς ελέγχους με ενδιαφέρον άκουσα την παρέμβασή σας αλλά είναι ένα θέμα που δεν είναι ακριβώς δικό μου θα μεταφερθεί και αυτό στον αρμόδιο Υπουργό. Τώρα, για το θέμα της εισαγγελία που είπατε, είναι κάτι που θα απαντήσω του Ευρωπαίου Εισαγγελέα που ετέθη, απήντησα βέβαια και στην ε, Επιτροπή ε, πριν από λίγο. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι ο Ευρωπαίος εισαγγελέα θα βοηθήσει πάρα πολύ στην πάταξη των ε, εγκλημάτων και ειδικά της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Είναι ένας θεσμός ο οποίος κατά την ε, άποψή μας είναι θετικός και πρέπει να προχωρήσει. Αναγνωρίζουμε όμως τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε κράτο μέλος λόγω των συνταγματικών διατάξεων που έχουν σχέση με την ε, ε, ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια και τη διάκριση των εξουσιών νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής και στο πώς ποια θα είναι η δομή αυτής της εισαγγελίας το ΜΕΝ και η εξάρτησή της με τους ε, εγχώριους εισαγγελίε των κρατών μελών. Άρα πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες και βεβαίως τι είδους ιεράρχησης θα υπάρχει. Η ίδρυση όμως της Ευρωπαϊκής Εγγυητικής Αρχής δεν πρόκειται να θίξει τον σκληρό πυρήνα των εθνικών αρμοδιοτήτων της εισαγγελικής αρχής εκάστου κράτους μέλους, αλλά αντιθέτως πρόκειται να ενδυναμώσει και να συσφίξει την ε, περαιτέρω συνεργασία των εθνικών εισαγγελικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κοινού σκοπού της ολοκληρωμένης προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια υπάρχουν μεγάλες ε, αρκετές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ να μην σα κουράσουν ειδικά θέματα, η αρχή τη επικουρικότητα κλπ. η οποία άλλε χώρε τη δέχτηκαν, άλλε όχι. Αλλά πρέπει να σα πω ότι δεν αποκλείεται και μια ενισχυμένη συνεργασία κατά το τέλο τη Προεδρία. Αυτό θα δούμε πώ θα πάνε οι εργασίε. Πάντως, ε, εν κατακλείδη σας λέω ότι είναι ένα ε, θετικό, ε, μια θετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωση γενικότερα και πρέπει να προχωρήσει. Τώρα, ε, είχαμε άλλο θέμα, νομίζω, για την νομοθετική πρόταση για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των ε, εισηγμένων ανωνύμων εταιρεών και αυτό είναι άλλων αρυπογείων αρμοδιότητα. Πάντως μπορώ να σας πω, ε, λόγω της παλιάς μου ιδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί και την Ελλάδα και πρέπει να μας απασχολήσει για το ζήτημα αυτό. Θα το συζητήσω και αυτό με τον κύριο Μιχελάκη και θα δω πώς μπορείτε να έχετε μία απάντηση ε, πιο έγκαιρη. Έχω προσωπική άποψη, αλλά νομίζω είναι κατάλληλο να σας ε, το πει ο ίδιος. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι διάκεμε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να σας πω ότι, αν επιτρέπετε τώρα, βέβαια είναι εκτός, όχι ως Προεδρία της ε, Ένωσης, αλλά Πήραμε πάρα πολλά μέτρα στην Ελλάδα για το ζήτημα, για παρόμοια ζητήματα και τελευταία ε, δημιουργήσαμε ε, και πάρα πολλούς ε, συμβουλευτικούς σταθμούς προστασίας των γυναικών μέσα για να προστατεύονται από πράξεις βίας. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς σταθμούς τέτοιους στην Ελλάδα. Και στην, υπάρχει και ένα σωματείο οργάνωση που έχει το όνομα της Σκούρα είναι μια, η πρώτη Έλληνα βουλευτή η οποία έγινε, που ασχολείται με ζητήματα τέτοια και μάλιστα θέλει να, να υπάρχει, συζητάνε και μέχρι και ποσόστοση ακόμα των γυναικών και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά υποχρεωτική ποσόστοση, αλλά και στην αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά και σε άλλες μορφές της γενικότερης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Ευχαριστώ πολύ. Er σας ευχαριστώ κύριε Ρέγνερ. Εσείς μια παρέμβαση πάλι. Όχι, είχα σκεφτεί το θέμα στα διοικητικά συμβούλια των γυναικών ποια αντιμετώπιση θα, αντιμετώπιση τύχαν, αλλά καλύφθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ που προσήλθατε. Ευχόμαστε στην Ελληνική Προεδρία κάθε επιτυχία και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας στους επόμενους μήνες σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία να σας συρρήξουμε. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και την Επιτροπή σας. Είμαστε σίγουροι ότι θα μας ε, συνδράμετε όπως εξάλλου έχετε κάνει και με τις προηγούμενες προεδρίες αλλά και τις πρώτες επαφές που έχουμε και έτσι με περισσότερη αισιοδοξία προσβλέπουμε στη βοήθεια σας πολύ περισσότερο που την έχουμε ανάγκη λόγω της μικρής διάρκειας που θα διαρκέσει εν ώψη των ε, ευρωεκλογών. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στην ημερήσια διάταξη δεν απομένουν πια τόσα πολλά. Έχουμε και την, το σημείο της κυρίας Στάιν, επικουρικότητα. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε ήδη επισημαίνω την γνωμοδότηση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Γερμανίας για τα διάφορα. Υπάρχουν παρατηρήσεις, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για τα διάφορα. Προσεχή συνεδρίαση, επόμενη συνεδρίαση, 10 Φεβρουαρίου στις 3 το απόγευμα, 15.00 εδώ στις Βρυξέλλες. Λίγη συνεδρίασή μας, σας ευχαριστώ, γεια σας.